Señor o presidente. Καλησπέρα σας, λέει ο κύριος ε, Σίλβα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έναρξη της συνεδριάσεως και πάλι και ας προχωρήσουμε στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Πρόκειται για την πρώτη δέσμη που αφορά την τροποποίηση τη συντονισμένη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη πανδημία COVID-19 για τον συνεπειών τη. Τα αποτελέσματα έχουν ω εξή. Τροπολογία υπαριθμών 2 εγκρίθηκε. Μπορεί να δείτε στην οθόνη τα αποτελέσματα και τον αριθμό των ε, ψήφων. Οπότε εγκρίθηκε έτσι το, η τροπολογία υπαριθμών 2 του κοινού.